πολύ προσεκτικά. Και όπω το είπε και η Προεδρία, θα λάβουμε υπόψη αυτό το οποίο είπατε και θα τα πούμε αυτά την Παρασκευή στο Συμβούλιο των Υπουργών. Euh, Ευχαριστώ κυρία Μάλστρομ. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση και η ψηφοφορία, όπως θυμήσατε και εσείς, θα γίνει στη μήνυ σύνοδο του Μαΐου. Σύμφωνα με τη μέση διάταξη ακολουθούν δηλώσεις Συμβουλίου και της Επιτροπής για τις καταστάσεις με τα νόματα των επιφατών PNR. Ο κύριος Λόπες Γκάριδο έχει το λόγο εξ του Συμβουλίου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας, η Προεδρία του Συμβουλίου υπέβαλε στο Κοινοβούλιο δύο συμφωνίες για τη χρήση ε, των καταστάσεων με τα νόματα των επιβατών. Είναι οι λεγόμενες συμφωνίες PNA του 2007, συμφωνία με τη ΣΥΠΑ και 2008 με, τις, με την Αυστραλία. Και ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, εγκρίνει και τις δύο συμφωνίες για να τεθούν οριστικά σε ισχύ, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζετε, είναι μεταβατικές απλώς και προσωρινές συμφωνίες αυτές εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα σύμφωνα με τη συνθήκη της Λαβώνας να αποφασίσει εάν εγκρίνει ή όχι τις συμφωνίες αυτές που ορίζουν τις συνθήκες ε, κάτω από τις οποίες μπορούμε με τρίτες χώρες να μοιραζόμαστε τις καταστάσεις των επιβατών ε, που ε, πετούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις χώρες αυτές. Το Συμβούλιο κατανοεί τα μελήματα και τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου Άλλωστε και προηγουμένως αυτά λέγαμε. Ακριβώς για τη συλλογή και τη συγκέντρωση αυτών των στοιχείων, των προσωπικών δεδομένων. Ας πούμε το γεγονός ότι ένα πρόσωπο επιβαίνει σε κάποιο αεροσκάφος. Για να φύγει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν το Συμβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει ένα γενικό έγγραφο προσανατολισμών ε, σχετικά. Οφείλω να σας πω ότι το σχέδιο ψηφίσματος που είδαμε μας φαίνεται πάρα πολύ καλό, μας ικανοποιεί η επικοδομητική στάση Βέβαια, αυτή τη στιγμή δεν ε, μπορείτε να ψηφίσετε, αλλά το σχέδιο ψηφίσματος, έλεγα, ε, ζητεί να δημιουργηθεί ένας κατάλληλος μηχανισμός για την αναθεώρηση των συμφωνιών. Στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι γεγονός ε, ότι υπάρχει μια έκθεση για την αναθεώρηση και όταν καταθέσει τη στάση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη νέα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε θα ε, γίνει γνωστή και η θέση του Συμβουλίου. Καθώς επίσης δεν υπήρξε και θεώρηση ούτε ε, για τη συμφωνία με την Αυστραλία, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει αν περιμένει ε, να έρθει πρώτα η αναθεώρηση της συμφωνίας και στη συνέχεια να αρχίσει μια νέα διαπραγματευτική εντολή. Ή όχι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα κάνει την πρότασή τη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο θα τη μελετήσει αναλόγω, Λαμβάνοντα πάντα υπόψη τι επιθυμίε και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τι ζητεί τώρα το Συμβούλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια ευρύτερη ρύθμιση, μια γενικότερη ρύθμιση για τη διαβίβαση αυτών των στοιχείων και δεδομένων των επιβατών. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι το 2007 είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια απόφαση πλαίσιο. Κατά τη διάρκεια όμως της Σουηδικής Προεδρίας εγκρίθηκε μια απόφαση που ήταν να διακοπεί η κάθε συζήτηση για την απόφαση πλαίσιο. Γιατί θεώρησε και σωστά η ε, Σουηδική Προεδρία ότι θα τεθεί σε ισχύ ε, η συνθήκη της Λισαβόνας και θα μπει στη συναπόφαση το θέμα αυτό, οπότε πρέπει να έχει λόγο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τότε η Προεδρία η Σουηδική το πάγωσε αυτό το θέμα. και ε, δεν ε, μπόρεσε να ληφθεί καμία απόφαση μέχρι την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, με τη διαδικασία της συναπόφασης. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει τεθεί σε ισχύ η σύνθηξη της Λισαβόνας. Εμείς ευθυγραμμιζόμαστε με τα όσα ζητάει το Κοινοβούλιο. Προς το παρόν δεν έχετε ψήφισμα, έχετε μόνο σχέδιο ψηφίσματος. Τρία είναι τα βασικά στοιχεία που θα ήθελα να υπογραμμίσω. Πρώτον, οι καταστάσεις και τα στοιχεία αυτά να χρησιμοποιούνται μόνο για το στόχο για τον οποίο ζητήθηκαν και δόθηκαν, αντίστοιχα με τα όσα συζητήσαμε προηγουμένως για το SWIFT. Δεύτερον, η συλλογή των στοιχείων αυτών θα πρέπει να συμφωνεί με τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και επιπλέον να υπάρχουν εγγυήσεις και ασφαλιστικές δικλείδες για τη διαβίβαση των στοιχείων αυτών σε τρίτες χώρες. Αυτές είναι οι τρεις βασικές σημαντικές αρχές, είναι στο σχέδιο ψηφίσματος και συμφωνούμε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Λόπεζ Γκαρίδο. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μάλστρομ για την Κομισιόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου. Η σημασία των στοιχείων PNR αναγνωρίζεται λένε και από περισσότερε χώρε, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, όσον αφορά την καταπολέμηση τρομοκρατία και άλλων σοβαρών εγκλημάτων. Για να διασφαλίσουμε τη σεβασμό των βασικών αρχών σεβασμού των ε, μάλλον προστασία των, ε, των ε, στοιχείων. Έχουμε ε, συμφωνίες με τη ΣΥΠΑ και με την Αυστραλία και τις έχετε ενώπιόν σας σήμερα για να τις εγκρίνετε. Ε, προτείνονται μια σειρά απαιτήσεων για όλε τι συμφωνίε PNR με τρίτε χώρε. Επίση, ε, ζητάτε από την Κομισιόν να διαπραγματευτείτε εκ νέου αυτέ τι οδηγίε αυτές μάλλον τις συμφωνίες, νομίζω πως είναι σοφή αυτή η στρατηγική. Στο ψήφισμα σας επίσης αναφέρεστε στην ε, συμφωνία PNR με τον Καναδά. Αυτή η συμφωνία συνδεόταν με διάφορες υποχρεώσεις ε, PNR. Τα έγγραφα αυτά ε, ξέπνευσαν στις 22 Σεπτεμβρίου του περασμένου χρόνου, πέρσι. Και εμεί ξαναδιαπραγματευτήκαμε με τον Καναδά. Για πρακτικού λόγου δεν κατέστη δυνατόν να γίνει αυτό πριν από το Σεπτέμβριο του 2009. Ωστόσο, αυτό δεν μειώνει το επίπεδο προστασία ε, στοιχείων ε, PNR που μεταφέρονται, που διαβάζονται στον Καναδά. Δεν υπάρχει ημερομηνία εκπνοή, δεν έχει ποτέ ε, πάυση ισχύ τη, άρα εξακολουθεί να ισχύει και το αρμόδιο Καναδικό Συμβούλιο έχει διαβιβάσει σχετική επιστολή προ την Κομισιόν και το Συμβούλιο ότι η δέσμευσή του παραμένει ε, η ίδια μέχρι ότου συναυθεί νέα συμφωνία. Να ευχαριστήσω τώρα την, την ε, εισηγήτρια κυρία Σόφια Εντεβέλτε για την επικοδομητική της στάση. Οι συμφωνίε με τις ΗΠΑ και την Αυστραλία παραμένουν εφαρμοστέ μέχρι ότου εγκριθούν οι νέε προτείνουμε ένα πακέτο PNR το οποίο θα αποτελείται βασικά από μια ε, επικοινωνία για μια σφαιρική στρατηγική PNR ε, με βάση τις γενικές ε, απαιτήσεις που, που περιλαμβάνει οποιαδήποτε συμφωνία PNR με τρίτες χώρες. Επίσης, οι οδηγίες αυτές θα ληφθούν υπόψη για τη ΣΥΠΑ, για την Αυστραλία αλλά και για τη νέα συμφωνία με τον Καναδά. Βασιζόμαστε σε μια αξιολόγηση επιπτώσεων και το πακέτο αυτό θα λάβει υπόψη τις συστάσεις όπως αυτές παρουσιάζονται σε αυτό το ψήφισμα αλλά και στο ψήφισμα του Νοεμβρίου 2008. Επιπλέον θα λάβει υπόψη τις συμβουλές του, επόπτη, του Ευρωπαίου Επόπτη για την προστασία δεδομένων και την άποψη των Εθνικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων. θα πρέπει να διατηρηθεί η συνέπεια ανάμεσα στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική PNR της Ένωσης. Ε, ε, καλωσορίζουμε λοιπόν αυτά τα συμπεράσματα και θα ενεργήσουμε σύμφωνα με αυτές τις ε, συστάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και τώρα το λόγο θα λάβουν οι ομιλητές εξ ονόματος των ομάδων και θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Άξελ Βόση για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη κυρία Επίτροπε, κύριε Προεδρεύον τα ίδια με το SWIFT και στο PNR. Καταβάλλεται ε, με ΑΙ μια προσπάθεια ε, εξισορρόπησης. Από τη μια έχουμε την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, από την άλλη έχουμε την ιδιωτική σφαίρα του καθενός και την αυτοδιάθεση της πληροφορίας ε, σχετικά με το άτομο του καθενός. αλλά δεν μπορεί να υπάρξει στην ψηφιακή εποχή εγγύηση χωρίς πληροφορία. Θα πρέπει ε, να δούμε πού ε, θα βρίσκεται το επίπεδο προστασίας και της ιδιωτικής ζωής και της πληροφορίας ε, για ε, τους πολίτες και του δικαιώματος να διαχειρίζονται οι ίδιοι αυτές τις πληροφορίες. Χρειάζεται μια πολύ λεπτή διάκριση εκεί. Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι χρειάζονται έλεγχοι, ε, προσφυγές, περιορισμοί για το χρόνο τήρηση των στοιχείων η λεγόμενη μέθοδος που θα πρέπει να ελεγχθεί αν μπορεί να επιτρέπεται σε έκτακτες περιστάσεις όλες οι διάζουσες και αν εκεί μπορούμε να βάλουμε και τη βαριά εγκληματικότητα, τα σοβαρά ε, ε, δικήματα όπως είναι παιδική ε, πορνογραφία, βιασμός, δολοφονία, λαθρεμπόριο ναρκωτικών, δουλεμπόριο γιατί και αυτά είναι θέματα προστασίας ε, της προσωπικότητας ε, και της αξιοπρέπειας των ατόμων. Θα πρέπει να αναβάλουμε τώρα την απόφαση, να ε, φτιάξουμε ένα μοντέλο βασικό για όλες τις επόμενες συμφωνίες και να δώσουμε εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα συμπεριλάβει όλα αυτά και στην προστασία των δεδομένων. Ενδεχομένως στο μέλλον να βρεθεί και κάποιος χώρος να σκεφτούμε τι κάνουμε για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της εγκληματικότητας σε συνεργασία ε, με τους ε, εταίρους μας στις Ηνωμένε Πολιτείες σε κάποιον κοινό οργανισμό γιατί ε, είναι παγκοσμιοποιημένη πλέον η εγκληματικότητα και χρειάζεται και παγκόσμια αντιμετώπιση. Ευχαριστώ. Η κυρία Σίπελ έχει τώρα το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω μερικά βασικά πράγματα για το θέμα αυτό. Βεβαίως υπάρχουν κοινά στοιχεία με το SWIFT αλλά και διαφορές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα αν ήταν υποχρεωμένο να ψηφίσει για τις καταστάσεις αυτές με τα ονόματα των επιβατών, δεν θα μπορούσε παρά να απορρίψει τη συμφωνία αυτή, γιατί παραμένουν σημαντικές και μεγάλες οι αμφιβολίες και θα έρθω στη συνέχεια λεπτομέρειες. Γι' αυτό δεν χάρηκα όταν έγινε λόγος για αναβολή της ψηφοφορίας. Σε αντίθεση με το SWIFT, ε, έχουμε κάθε λόγο να αναβάλουμε. Βέβαια δεν λέω να αναβληθεί επαόριστον η ψηφοφορία και να διαιωνίζεται μια μεταβατική προσωνή συμφωνία για χρόνια ολόκληρα. Όχι. Θέλουμε το συντομότερο να υπάρξει νέα διαπραγματευτική εντολή ή δυνατόν πριν τις ενές διακοπές για να επικρατήσει σαφήνεια πάρα πολύ γρήγορα και στις λεπτομέρειες. Τι κάνουμε με τα στοιχεία αυτά, τι στοιχεία στέλνουμε και πώς. Η προστασία των δεδομένων ε, παίζει σημαντικό ρόλο και θα ήθελα εδώ να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία που έχω για να μπω και στις λεπτομέρειες. Ποια στοιχεία στέλνουμε. 19 ε, μεμονωμένα ε, δεδομένα είναι αυτά. Είχα συζητήσει και επαφέ και μου εξήγησαν ότι αν θέλει κάποιο, από αυτά τα 19 στοιχεία μπορεί να καταλάβει ποιος είναι ο άνθρωπος, να βρει το προφίλ του. Δεν έχουμε εμεί συμφέρον να συμβεί κάτι τέτοιο, μα λένε. Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα, μετά τα σβήνουμε τα στοιχεία. Ωραία. Αλλά εάν ε, τόσα πολλά στοιχεία ε, χρησιμοποιηθούν στρεβλά και μπορεί κανείς να ταυτοποιήσει το πρόσωπο, αναρωτιόμαστε είναι σωστό, επιτρέπεται να συλλέγονται καν και να διαβιβάζονται. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό ερώτημα. Και επίσης στα στοιχεία που διαβιβάζονται πρέπει να ξέρουμε τι ισχύει για την προστασία τους. Ξέρουμε ήδη ότι στις δύο συμφωνίες με ΙΠΑ και Αυστραλία οι ε, διατάξεις είναι πολύ διαφορετικές ε, σε ό,τι αφορά αιτήσει άλλων ε, χωρών που θέλουν να συνάψουν και αυτές τις αντίστοιχε συμφωνίες. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αν συμφωνήσουμε πάντα αυτό θα πρέπει να είναι πολύ αυστηρό. Επίσης, για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται αυτά τα δεδομένα. Πάρα πολύ Λεπτομερή ρύθμιση χρειάζεται. Στην αρχή μα λένε κατά πολέμηση τη τρομοκρατία, μα είπανε. Α, τώρα το έχουν περάσει και στα σοβαρά εγκλήματα. Ωραία, να το συζητήσουμε αυτό. Αλλά να μπούμε σε λεπτομέρειε και με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Ήδη γνωρίζουμε ότι στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ο πολιτισμό ο από χώρα σε χώρα διαφέρει πάρα πολύ. Οπότε τι είναι σοβαρό έγκλημα ε, ή σοβαρά αδικήματα. Έτσι, εδώ χρειάζεται ρύθμιση λεπτομέρειες ότι βεβαίω και σε περίπτωση σοβαρή εγκληματικότητα θα πρέπει να διαβάζεται αυτό ο κατάλογο. Στο μέλλον λοιπόν στην εφαρμογή της συμφωνίας αυτής θα πρέπει να έχουμε και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο Προεδρεύων του Συμβουλίου είπε ότι έγινε μια πρώτη αναθεώρηση της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσημα τα αποτελέσματα δεν τα έχουμε ακόμα. Το Φεβρουάριο έγινε αυτό. Ε, θα επιθυμούσα ε, να μην έχουμε μόνο τακτικές εκθέσεις αλλά οι εκθέσεις αυτές να διαβιβάζονται το συντομότερο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό και σημαντικό να έχουμε ενιαία συμφωνία. Να ξανακοιτάξουμε αυτό το θέμα των δεδομένων, αλλά μέχρι τώρα έχω την εντύπωση ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στη σωστή κατεύθυνση για να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία και προσβλέπω σε αυτή. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Ινετ για τρει και μισή λεπτά. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνάδελφοι, ω εισηγήτρια θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους σκεώδει εισηγητέ για την εξαιρετική, ευχάριστη και πλήρη συνεργασία που κατέληξε σε ένα κοινό ψήφισμα. Και φυσικά αυτό, αυτή δεν είναι η τελευταία, φάση. Οι συζητήσει θα συνεχιστούν, οπότε σήμερα εξετάζουμε το αίτημα για, για συγκατάθεση από το Συμβούλιο για τι δύο συμφωνίε με τη ΣΥΠΑ και την Αυστραλία. Ε, το σώμα μας ανέκαθεν ήταν επικριτικό όσον αφορά τη χρήση και τη μεταφορά ε, ε, ποινικών ε, στοιχείων Μάλιστα το 2004 το Κοινοβούλιο ε, έλεγξε ενώπιον του δικαστηρίου τη συμφωνία πριν την υπογράψει με τη ΣΥΠΑ. Θα ήταν λάθος λοιπόν να, να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας χωρίς ε, να την μελετήσουμε εις βάθος. Ωστόσο συμφωνούμε πως αν απορρίψουμε τις δύο συμφωνίες θα δημιουργήσουμε νομική αβεβαιότητα για τους πολίτες και, τους, ε, και τις αεροπορικές εταιρείες. Γι' αυτό και ε, θέλουμε να κάνουμε την ε, ψηφοφορία επί τη βάση ενό σαφού συνόλου αρχών. Είμαι ευχαριστημένη γιατί το Συμβούλιο και η Επιτροπή επέλεξαν να δεχτούν αυτή την αρχή και έτσι μπορούμε να δουλέψουμε γρήγορα και με ευελιξία και να εγκρίνουμε το πακέτο πριν τις ε, θερινές διακοπές. Μια τέτοια προσέγγιση είναι πιο ρεαλιστική προσέγγιση γιατί όλα είναι και περισσότερες χώρες ζητούν την ε, μεταφορά των στοιχείων αυτών. Βέβαια υπάρχει το θέμα της συμφωνίας με τον Καναδά όποιο και αν είναι το νομικό της καθεστώς, που δεν είναι πολύ ξεκάθαρο, καθώς και η πρόταση για ένα νέο PNR. Αυτό το σχέδιο ψηφίσματος ορίζει διάφορες βασικές αρχές, ελάχιστες προδιαγραφές για το πακέτο PNR και υπάρχουν και διάφορες προϋποθέσεις για την συγκατάθεσή μας. Βασικά στοιχεία, βασική λέξη είναι η αναλογικότητα, διότι θα πρέπει να αποδειχτεί με πιστικό τρόπο ότι το ίδιο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί με λιγότερο διαιτητικά μέσα. Αυτό είναι το κλειδί για όλα. Πρέπει να εξετάσουμε τα στοιχεία ε, έστα και να διαχωρίσουμε σαφώς ανάμεσα στην μαζική μεταφο... συλλογή και χρήση στοιχείων όλων των επιβατών για το στόχο των ε, ερευνητών όπως το profiling και η εξόριξη στοιχείων και από την άλλη πλευρά στοχοθετημένες έρευνες για μη υπόπτους ε, για τον εντοπισμό δηλαδή ανθρώπων που επιβαίνουν σε μια πτήση. Πρέπει σε αυτά να γίνει, να γίνει σαφής διάκριση. Ε, Περιορισμό των στόχων λοιπόν, σύμφωνα με προηγούμενα ψηφίσματα και επιμένουμε τα στοιχεία να χρησιμοποιούνται μόνο για την επιβολή του νόμου και τη σκοπού ασφαλείας και με πολύ συγκεκριμένο ορισμό του τι είναι αυτό, οργανωμένο Διεθνέ έγκλημα και Διεθνή τρομοκρατία. Πρέπει να καταστήσουμε απόλυτα σαφέ για ποιο πράγμα μιλάμε. Οποιαδήποτε χρήση PNR θα πρέπει να συμφωνεί με τα στάνταρ Προστασία δεδομένων τη Ένωση. Είναι πρωταρχική μα ευθύνη να αντιπροσωπεύσουμε τα συμφέροντα όλων των Ευρωπαίων πολιτών πολιτών γιατί έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν πως στις διεθνείς σχέσεις και στις εσωτερικές μας πολιτικές ε, συμμορφωνόμαστε προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και τέλος θα πρέπει να παρέχουμε στις αρχές επιβολής του νόμου και ασφάλειας ε, τις απαραίτητες, τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να κάνουν τη δουλειά τους σωστά και έχουμε τη δυνατότητα να προστατεύουμε τις ελευθερίες μας και τα δικαιώματά μας. Νομίζω πως με το επόμενο πακέτο PNR έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να τα φτιάξουμε όλα αυτά σωστά. Ευχαριστώ κυρία Ιντιβέλτη, κυρία, ο κύριος Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν θέλω να επι... επαναλάβω αυτά που είπαν ε, πολύ σωστά οι συναδελφοί, αλλά να κάνω ο... Ο... γενικές παρατηρήσεις. Αν δεν έχετε δει την ταινία No to Report, ε, Minority Report, θα σας έλεγα να το δείτε. Διότι ε, υπάρχουν στοιχεία που συλλέγονται πριν υπάρξει ποινικό αδίκη και ε, υπάρχει το συνέστημα ότι ο άνθρωπος παρακολουθείται συνέχεια. Είναι ένα σύστημα το οποίο υποτίθεται ότι φροντίζει για την ασφάλεια και τελικά όλα καταραίουν. Δεν ε, θέλω να αναφερθώ περαιτέρω σε αυτή την κατάσταση αλλά η ε, επίθεση σε όλες τις σε όλα τα στοιχεία των επιβατών ε, ισχύει από τις 10 ε, Σεπτεμβρίου του 2001 στις Ηνωμένε Πολιτείες και αυτή η ανεξέλεγκτη ε, επίθεση βρίσκει σαν θύμα την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου προσκρούει σε, σε αντισυνταγματικότητα διότι υπάρχει αυθαιρεσία η ε, ανταλλαγή στοιχείων με τις Ηνωμένε Πολιτείες και την Αυστραλία είναι παραβίαση των δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων πράγμα το οποίο έχουμε πει επανειλημμένος οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ε, σαν ε, Συμβούλιο ούτε σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ζητάμε να υπάρξει ένα, μια κατάσταση κατάσταση πρώτων ποινικών ε, δικημάτων. Τώρα ο κύριος Ρίτσαρτ Καρνεύσκη για ε, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όπως και ο προλαβής σας, εγώ θα ήθελα να επισημάνω το γεγονό ότι θα ήταν ενδιαφέρον να μιλήσουμε για την τέχνη την έβδομη του σινεμά. Αλλά επανέρχομαι στα Passenger Name Records. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι έχει ένα χαρακτήρα αυτονόητο. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αυτό το θέμα το οποίο είναι αρκετά απλό και αυτονόητο έχει αποτελέσει αντικείμενο μια θεσμική αντιπαράθεσης μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Κατά την άποψή μας, το <clears throat> σχέδιο αυτό για τα PNR έχει μία βάση η οποία είναι ορθή, αλλά έχει παρουσιαστεί με έναν τρόπο αυθαίρετο από το Συμβούλιο χωρίς την απαραίτητη διαβούλευση με το Κοινοβούλιο. Και επομένως το αποτέλεσμα ήταν μια αποτυχία. Ακόμα και αυτοί λοιπόν οι οποίοι θα θέλανε καταρχήν να υπάρχουν ε, αυτά τα στοιχεία τα οποία θα δίδονται στι Αμερικανικέ Αρχέ έχουν αντίρρηση σήμερα γιατί θέλουν να διατηρήσουν τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου ως ενό ισχυρού θεσμικού οργάνου. Και με αυτόν τον τρόπο πάρα πολλοί έχουν βρεθεί ξαφνικά στην, ε, στην χωρία των αντιπάλων του, της ρύθμισης αυτή, αυτής λόγω της τάσης του Συμβουλίου. Αν φτάνει λοιπόν αυτό, υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος αυτών οι οποίοι υποστηρίζουν να δοθούν αυτά τα ε, στοιχεία, θεωρούν ότι πρέπει να κατηγορήσουν, ότι πρέπει να καταγγείλουν μάλλον και να τιμωρήσουν το Συμβούλιο για την αλαζονία με την οποία έχει κάνει αυτά μαζί με τα ύδατα μπανίου έχει αποσταλεί από το παράθυρο και των πεδίων, όπως λέμε στην χώρα μου. Και έτσι δεν λοιπόν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία. Αντίθετα με τους προηγούμενους ομιλητές, θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την θετική μου αντιμετώπιση έναντι του κυρίου Άλμπρεκτ για την σύγκριση που έκανε με το σινεμά. Μερικές φορές είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε πολιτιστικά επιχειρήματα και είναι ενδιαφέρον να ασχολούμαστε και με τις κοινωνικές αλλαγές και εξελίξεις. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ινφέλτ, την ε, εισηγήτρια, για την προστασία της προσωπικής ακαιρεότητας και της ασφαλείας δικαίου, που ήταν η κύρια Μεριμνάτης. της. η Ισπανική Προεδρία είπε ότι η αεροπορία είναι ο τρόπο με τον οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί η ελευθερία διακίνηση, ένα θεμελιώδε ανθρώπινο δικαίωμα. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μα όταν λέμε για τα PNR. Γιατί αυτά τα μητρώα, τα PNR, μπορούν να εμποδίσουν ορισμένα άτομα από το να χρησιμοποιήσουν αεροπορικέ πτήσει. Αυτό επηρεάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, επηρεάζει την ελευθερία τη διακίνηση των ατόμων και προφανώς αυτό επηρεάζει την εφαρμογή διεθνών συνθήκων σε σχέση με τα δικαιώματα των πολιτών μας. Νομίζω ότι ο στόχος που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσει δηλαδή την ελευθερία διακίνησης των πολιτών είναι καταρχήν να εξαλείψει τα εσωτερικά σύνορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να βελτιώσει την διακίνηση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε ότι αυτό όμως δεν συμβαίνει για αυτούς οι οποίοι αιτούνται ασύλου, για τους πρόσφυγες και άλλα άτομα. Πολλέ φορέ αυτά τα άτομα, οι αιτούντε άσυλο και οι πρόσφυγε, είναι απλώ γυναίκε και παιδιά που δεν έχουν πραγματικέ δυνατότητε. και το να αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν μπορούν να πετάξουν ή όχι είναι μερικέ φορέ θέμα ζωή και θανάτου για τα άτομα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γι' αυτό το λόγο εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την πλευρά τη ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσέξουμε πάρα πολύ για το πώ θα χρησιμοποιηθούν τα PNR στη συνέχεια. Αυτό που μα ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να εξασφαλίσουμε την ελευθερία διακίνησης αλλά και τον σεβασμό των διεθνών συμβάσεων και των δικαιωμάτων των πολιτών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μέλτσερ δεν είναι παρόν. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπούσου Τιλ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για το SWIFT είχαμε πει ότι υπήρχαν μια σειρά από προϋποθέσεις για να μπορέσει να λειτουργήσει μια τέτοια συμφωνία. Και αυτό είναι πραγματικά ένα δίδαγμα για το Συμβούλιο. Εφόσον έχουμε περισσότερες εξουσίες ως Κοινοβούλιο, έχουμε και περισσότερες ευθύνες και πρέπει να τις ασκήσουμε. Και επομένως η στρατηγική που ακολουθεί το Κοινοβούλιο για τα PNR δείχνει ότι ακόμα και το Κοινοβούλιο έχει κατανοήσει ότι έχει αυξημένες ευθύνες. Είναι λοιπόν μια πολύ θετική υπογράμμιση αυτή. Ένα δεύτερο σχόλιο τώρα. Η συμφωνία αυτή είναι τόσο σημαντική. Κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντική. Γιατί ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας είναι ένας σημαντικός αγώνας για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών και επομένως έχουμε μια μεγάλη ευθύνη για τους πολίτες μας που την επομιζόμαστε. Αν συμβεί κάτι, εμεί θα είμαστε υπόλογοι απέναντι στου πολίτε μα. Θα μα ρωτήσουν τι έχετε κάνει για να εξασφαλίσετε την ασφάλειά μα. Τρίτο σημείο. Αυτή η συμφωνία θέτει θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ιδιωτική ζωή των πολιτών. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι πράγματι θέτει τέτοια ζητήματα, οδηγεί σε κάποιε ανησυχίε για του πολίτε μα, γι' αυτό είναι απαραίτητο να το εξετάσουμε το θέμα αυτό και να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία η οποία διασφαλίζει τα συμφέροντα τα θεμητά συμφέροντα των πολιτών μας για την ιδιωτική του ζωή. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ένα ορθό ψήφισμα σε σχέση με το περιεχόμενό του, ένα ισορροπημένο ψήφισμα και καταδεικνύει σαφώς τι θέλει να κάνει το Κοινοβούλιο και τι επιζητεί. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να δείξουμε σε όλους ότι εμείς χρησιμοποιούμε τις εξουσίες μας με ένα υπεύθυνο τρόπο. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ την εισηγήτρια για τη θαυμάσια εργασία της στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Μπουσουτήλ. Ευχαριστώ. Ο Σαΐντ Ελκαντράουι για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, η συζήτηση αυτή μας υπενθυμίζει α, τη συζήτηση που κάναμε προηγουμένως για το SWIFT. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και στην προστασία της ε, ιδιωτικής σφαίρας, γιατί και τα δύο πράγματα είναι πολύ σημαντικά. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στις ενέργειες μεταφορές αυτές τις τελευταίες μέρες μας δείχνουν πως η μεταφορά ατόμων και εμπορευμάτων είναι πολύ σημαντική στην εποχή μας. Κάποια στιγμή όλοι μας παίρνουμε ένα αεροπλάνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε με μόνιμο τρόπο να μεταδίδουμε τα δεδομένα χωρίς να το σκεφτούμε και χωρίς να έχουμε καλές εγγυήσεις ότι θα χρησιμοποιηθούν σωστά αυτά τα δεδομένα. Οι Αμερικανικές αρχές εδώ και καιρό χρησιμοποιούν διάφορες πηγές πληροφοριών για να αντιληφθούν αν ένα άτομο είναι ύποπτο ή όχι και την, ε, τις θεωρήσεις και τη διαδικασία των θεωρήσεων τη χρησιμοποιούν και τη διαδικασία το, του check-in. Και πρόσφατα στην Ουάσιγκτον διαπίστωσα ότι 24 ώρες το 24ωρο υπάρχει μια ομάδα αμερικάνικη ε, που καταρτίζει ένα κατάλογο αφήξεων που ξεκινάει από 5.000 άτομα και μετά καταλήγει σε ένα short list ε, ατόμων που τους απαγορεύεται η επιβίβαση στις, προς την Αμερική. Επομένω, υπάρχουν εδώ κυρώσει για τα συγκεκριμένα άτομα. Γι' αυτό χρειάζονται κάποιε ελάχιστε εγγύησει, όπω αυτέ που αναφέρει το ψήφισμα για, τα, για όλα τα άτομα. Νομίζω ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε την διεθνή τρομοκρατία και τη διεθνή εγκληματικότητα, αλλά με τρόπο που να σέβεται ε, τις προϋποθέσεις ε, για την ε, ιδιωτικότητα και την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας. Υπάρχουν επίσης δεδομένα PNR που είναι όλους ιδιαίτερως ευαίσθητα. Και εδώ φοβάμαι ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι ανοιχτά σε διάφορες ερμηνείες. Εγώ προτείνω να βάλουμε μια ανωτελεία και να δώσουμε μια νέα εντολή. Περιμένω περισσότερες διευκρινήσεις και από το Συμβούλιο και από την Κομισιόν. Η κυρία Σαρτζεντίνη για 1,5 λεπτό έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κυρία Ιντβελτ παρουσίασε ένα θαυμάσιο ψήφισμα και συμφωνώ μαζί της ότι πρέπει να καταλήξουμε σε μία κοινή θέση για όλες τις συμφωνίες PNR ε, τις μελλοντικές. Πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια δεδομένα που για λόγους τρομοκρατίας πρέπει να μεταδίδονται, αλλά πρέπει να είναι μειωμένος ο αριθμός τους. Και αυτά τα δεδομένα πρέπει να χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο σκοπό. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο λόγο και δεν μπορούν να αποθηκεύονται για έναν αόριστο, για ένα αόριστο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε έμφαση στο, στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η συνθήκη για τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων έχει υιοθετηθεί και θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας. Και πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας και για τη διαβίβαση των δεδομένων PNR. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να επιφορτιστεί με το θέμα αυτό του PNR. Η Κομισιόν πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη. Επίσης κάτι άλλο που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι το εξή. οι πολίτες έρχονται σε επαφή με τις αμερικάνικες εταιρείες μέσω μιας ε, εταιρείας που είναι εταιρεία εναέριων μεταφορών στις περισσότερες περιπτώσεις ε, και ποτέ δεν θα έπρεπε αυτή η εταιρεία να παίξει το ρόλο του ενδιάμεσου. Η κυρία Έρνστ για ένα λεπτό έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, Υπάρχουν διάφορα τραγούδια και μιλάνε για μια γιορτή πάνω από τα σύννεφα, αλλά εδώ κάπου πρέπει να τελειώσει αυτή η γιορτή. Διότι υπάρχουν ήδη περιορισμοί των ελευθεριών και γι' αυτό το είδε και ένας συνάδελφος τον Αύγουστο και ε, το αεροπλάνο στο οποίο βρισκόταν ε, δεν έλαβε άδεια να ε, διέλθει από τους Αμερικανικούς εθέρες. Ε, και πρόκειτο για ένα λάθος, διότι υπάρχουν διάφορα στοιχεία τα οποία διαβιβάζονται, πιστοτικές κράρτες, στοιχεία διαβατηρίου, χωρίς να υπάρχει πραγματική προστασία δεδομένων. Και θέλω να σας πω ότι και αυτό απορρίπτουμε και μία σειρά από δεδομένα τα οποία καλύπτονται από την ονομασία PNR. Γι' αυτό και δεν θα στηρίξουμε την πρόταση αυτή υπό την τωρινή της διατύπωση διότι ε, δεν είναι σωστή. Θα ήθελα να σας πω τελικά ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε να ε, υπάρξουν ε, περαιτέρω τέτοιες ρυθμίσεις και δεν είναι δυνατόν να δίνουμε τα στοιχεία των Ευρωπαίων πολιτών στη ΣΥΠΑ διότι θα έπρεπε και αυτά μας δίνουν τα δικά τους. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μάνφρετ Ρούμπερ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε. Ε, Βέμπερ. Ευχαριστώ. Καταρχήν και εγώ θα ήθελα να κάνω μία σύγκριση με, στη συζήτηση SWIFT διότι βλέπω ότι το ε, Συμβούλιο είναι πολύ δεσμευμένο στο θέμα αυτό. Μιλάμε για τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, και βλέπουμε πώς αυτή επηρεάζει το Συμβούλιο ο οποίος θέλει να προασπίσει περαιτέρω τους πολίτες οπότε ελπίζω το ίδιο θέλει να κάνει και με τη διαβίβαση των και να προασπίσει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι όλοι συμφωνούμε ότι από πλευράς νομικής ασφαλείας για τις αεροπορικές εταιρείες αυτές οι συμφωνίες έχουν ίσως κάποιο νόημα αλλά νομίζω ότι έχουμε σωστά διατυπώσει ποιες είναι οι προδιαγραφές τις οποίες απαιτούμε. Και θα ήθελα επίσης να αναφέρω ένα άλλο θέμα το οποίο δεν έχει άμεση σχέση με τη συνθήκες αλλά με τη συζήτηση ε, με το Συμβούλιο. Δηλαδή αν χρειαζόμαστε και ένα ευρωπαϊκό ότι ε, ε, είχαμε την περίπτωση του Ντιτρόιτ που ήταν η μεγαλύτερη απειλή πέρυσι πριν τα Χριστούγεννα. Διαπιστώσαμε λοιπόν τότε ότι στη Μεγάλη Βρετανία γνώριζαν ότι ήταν επικίνδυνο το άτομο αυτό. Αλλά αυτοί οι οποίοι αποφάσισαν αν θα επιβασίσει στο αεροπλάνο ή όχι δεν είχαν τα στοιχεία αυτά. Δηλαδή πιστεύω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, ε, ότι δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι επικίνδυνοι, αλλά το θέμα είναι τα στοιχεία να μεταβιβάζονται εκεί που τα χρειαζόμαστε πραγματικά. Διότι στο Τολέδο η Ισπανική Προεδρία είχε δεσμευτεί και την ευχαριστώ για αυτό ότι θα ενισχύσει την ε, αντιτρομοκρατία στην Ευρώπη και τον αγώνα της πράγμα όμως το οποίο ε, ε, δεν υιοθετήθηκε από τους υπουργούς αντιθέτως ζητούν να συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία και νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο εύκολο ε, το θέμα αυτό για τους υπουργούς εσωτερικών θα ήθελα λοιπόν καλύτερα να στηρίξουν την, το έργο των αρχών θα ήταν πολύ καλύτερο το λόγο έχει η κυρία Τάνια Φασόν για τρία λεφτά Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι πεπισμένη ότι όλοι οι ευρωβουλευτές γνωρίζουν τη σημασία των ακριβών πληροφοριών για την εξασφάλιση της ελευθερίας, της ασφάλισης συγγνώμη, ε, στις ε, μεταφορές μας. Και το χάος της εναέριες μεταφορές ε, δείχνει ακριβώς το μεγάλο αριθμό των επιβατών καθημερινά. Υπάρχουν τώρα ε, μάζες ολόκληρες επιβατών που περιμένουν στην ουρά για μια θέση στο πρώτερο πλάνο που θα απογειωθεί. Η διαβίβαση δεδομένων στις αρχές για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ε, είναι απόλυτα θεμητό αίτημα. Δεν μπορώ να αντιταχθώ στη χρήση αυτών των δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι στις συμφωνίες PNR δεν έχουμε μία δέσμη κριτηρίων για τα δεδομένα που θα πρέπει να διαβιβαστούν. Και δεν γνωρίζουμε και τους στόχους. Γιατί διαβιβάζονται αυτά τα δεδομένα και πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα. Υποθέτω ότι θα υπάρξει μια εντολή για αυτή τη συμφωνία, ε, μάλιστα πριν από το καλοκαίρι. Ίσως οι συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις μεμονωμένες χώρες θα είναι ιδίου επίπεδου με ίδιο επίπεδο προστασίας ε, των δεδομένων και ασφάλειας. Τι μέτρα θα χρησιμοποιηθούν, ούτω ώστε να εμποδίσουμε τη χρήση των δεδομένων PNR για λάθος σκοπούς. Γιατί ε, το προφίλ των ατόμων με βάση το τη φυλή τους, την, υγεία, την ηλικία τους, το σεξουαλικό τους προσανατολισμό κτλ. Αυτό είναι απαράδεκτο. Επίσης, τα συστήματα συλλογής των δεδομένων ε, είναι διάτρητα. Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε την διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών χωρίς σωστή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των αντικρομοκρατικών οργανώσεων. Το θυμηθήκαμε αυτό ε, με την πρόσφατη απόπειρα που έγινε ε, στη πτήση για τον Detroit. Ο στόχος είναι η καλύτερη συνεργασία και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Σύμφωνοι. Δεν μπορώ να πω όχι σε αυτή τη συμφωνία, γιατί αυτή η συμφωνία εξασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών μας. Αλλά σωστό είναι επίσης ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν παρεμβάσεις και σφετερισμοί των δικαιωμάτων των πολιτών. Ε, η κυρία Λίχτενμπέργκερ. Είναι το δεύτερο θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε που έχει να κάνει με μια συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείε, το οποίο συνάπτεται με πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αυτό ουσιαστικά υπογραμμίζει την πρόταση του αρμοδίου για την προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων ότι θα είχε νόημα να υπάρχει καταρχήν μια διατλαντική συμφωνία πλαίσιο σε σχέση με την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων. Νομίζω θα ήταν λογικό και από τις δύο πλευρές και θα μας ελάφρωνε πάρα πολύ από το άκθος αυτών των συζητήσεων. Είναι γεγονός ότι από τη μία πλευρά πρέπει να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να σκεφτούμε και την προστασία των δεδομένων ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορεί η, η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απλώς να υιοθετεί μηχανιστικά αυτά τα οποία προτείνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο να μπορεί να βρίσκεται σε επίπεδο ισότητα με τι Ηνωμένε Πολιτείε και να μπορεί να χρησιμοποιήσει και τα δικά μα πρότυπα για την προστασία των δεδομένων, τα οποία θα πρέπει να είναι αντι, αντικείμενο ε, συζήτηση και διαπραγματευσή. Το τι είναι αδίκημα λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα συμφωνία και των δύο πλευρών. Εάν δεν υπάρξει επιπλέον η προστασία των δεδομένων, από τη δική μας πλευρά είναι όχι για τη συμφωνία αυτή. Δεν μπορούμε να τη δεχτούμε. Ο κύριο Κάρδο Κουέλιου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ Λόπε Γκαρίδο, κυρία Επίτροπε Μάλστρομ, εμεί έχουμε εκφράσει ήδη την ανησυχία μα σε ό,τι αφορά τη μετάδοση των στοιχείων PNR προ τι ΗΠΑ. Αυτό είναι γεγονός ότι μετά από όλες τους ελέγχους που έχουν γίνει δεν θεωρούμε ότι υπάρχει η εξασφάλιση της προστασίας αυτών των δεδομένων. Οι συμφωνίε που είχαμε κάνει με την Αυστραλία και τον Καναδά είχαν το στοιχείο τη αμοιβαιότητα και εξασφάλιζαν το περιορισμένο στο χρόνο και στην έκταση της πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα, πάντα με δικαστικό έλεγχο. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρχουν γενικοί κανόνες οι οποίοι θα είναι το πλαίσιο με στο οποίο μπορούν να συναυθούν συμφωνίε αυτού του είδου με τρίτε χώρε. Και εξάλλου, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλέ τέτοιε αντίστοιχε αιτήσει από, από άλλες χώρες που έχουν πολύ πιο ανησυχητική παράδοση ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμεί λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη δημιουργία ενό ενιαίου συστήματο για την Ευρωπαϊκή Ένωση με πλήρη συμμετοχή τη Ευρωπόλ σε όλη αυτή τη διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπη για μένα, οποιαδήποτε συμφωνία θα είναι μονάχα αποδεκτή μόνο αν έχει το απαραίτητο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δικαιωμάτων και θα υπόκειται στους τρέχοντες κοινοτικού κανόνες για την προστασία αυτών των δικαιωμάτων. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα τα οποία θα δώσουμε εμείς δεν θα μπορέσουν να δοθούν σε τρίτες οι οποίοι θα έχουν έτσι ένα αυτόματο δικαίωμα πρόσβαση στα προσωπικά μας δεδομένα. Εγώ υποστηρίζω λοιπόν την πρόταση της κυρίας Σινβέλτ που εκφράζει την άποψη των πολιτικών ομάδων και όλου του Κοινοβουλίου ότι είναι απαραίτητο να δοθεί περισσότερο χρόνο για να μπορέσουν να γίνουν διαπραγματεύσει και να καταλήξουμε έναν τρόπο ο οποίο ανταποκρίνεται στι ανησυχίε όλων των μελών του Κοινοβουλίου και όλων των ομιλητών οι οποίοι έλαβαν το λόγο. Κάτσε the τώρα. Η κυρία Τικάου έχει το λόγο. Ένα λεπτό κυρία Τικάου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ο προσωπικός χαρακτήρας των δεδομένων είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των πολιτών. Μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουν ενισχυθεί τα στοιχεία αυτά σε ό,τι αφορά τον ε, υποχρεωτικό χαρακτήρα της εφαρμογής της χάρτας θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οποιαδήποτε διαδικασία η οποία αφορά αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να βασίζεται στους κανονισμούς οι οποίοι διέπουν τα θέματα αυτά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί οποιαδήποτε διεθνή συμφωνία η οποία αφορά τα δεδομένα PNR θα πρέπει να γίνει δεκτή και μόνο εάν οι συνομιλητές μας αποδέχονται τις διατάξεις αυτές οι οποίες αναφέρονται στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αφορά την επικοινωνία με ευρυζωνικά μέσα την ε, διαδικασία αποθήκευσης και πρόσβασης στα δεδομένα. Οποιαδήποτε λοιπόν συμφωνία για τα PNR θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η αποθήκευση και η ε, επεξεργασία αυτών των δεδομένων θα γίνεται μονάχα σε εγκαταστάσεις οι οποίες προβλέπουν διασφαλίσεις ανάλογες με αυτές που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς λοιπόν θα έβλεπε αυτό το θέμα ο Ευρωπαίος πολίτης. Οπότε εφόσον δεν ε, υπάρχουν άλλοι ομιλητές θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου τον κύριο Λοπές Γαρίντο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σταθώ σε τρεις παρατηρήσεις υπομορφή συμπερασμάτων από τη μεριά του Συμβουλίου για αυτό το τμήμα της συζήτησης. Το πρώτο συμπέρασμα το ανέφερε ήδη ο κύριος Βέμπα ο οποίος μίλησε για την δυνατότητα να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό σύστημα PNR. Εμείς φυσικά θέλουμε να υπάρξει ένας κανονισμός για τα θέματα αυτά σε ό,τι αφορά την ε, μεταβίβαση στοιχείων επιβατών ιδιαίτερα στον ενάρι, στις εναέριες μεταφορές και από την άποψη αυτή ζητήσαμε πράγματι στην Κομισιόν να προβεί στην εκπόνηση μιας μελέτης για τα θέματα αυτά και εν καιρό να μας υποβάλει μια πρόταση κανονισμού για τα ζητήματα αυτά. Το ψήφισμα της κυρίας Ιντφέλτ λέει ότι υπάρχει μία μελέτη αντικτύπου που αφορά τον ενδεχόμενο αντίκτυπο που μπορεί να υπάρξει για την ιδιωτική ζωή των επιβατών. Εξετάζει δηλαδή σε ποιο βαθμό η αποτελεσματικότητα και η αναλογικότητα που είναι δύο βασικές αρχές που πρέπει να έχουμε πάντα στο πνεύμα μας έχουν αποτέλεσμα σε βάρος της ιδιωτικής ζωής των πολιτών. Δηλαδή μέχρι πού είναι το ερώτημα πρέπει να φτάσει το Σύνολο των Κανονιστικών Ρυθμίσεων στην ε, Ευρώπη για τα PNR και πώς θα προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα. Η κυρία Φαγιόν έθεσε το ερώτημα του ποια είναι τα κατάλληλα μέτρα τα οποία μπορούμε να αναλάβουμε. Νομίζω ότι μπορεί να μας διαφωτίσει εδώ και η συζήτηση που κάναμε προηγουμένως για το SWIFT. Νομίζω ότι οι βασικές αρχές για τις οποίες σύμφωνουμε και η ΜΕΝ και η ΔΕ θα πρέπει να πριτανεύσουν και στην τρέχουσα περίπτωση. Μιλάμε για τα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή, τα δικαιώματα να υπάρχει ακεραιότητα της προσωπικότητας και της εικόνας του κάθε ατόμου, αυτά είναι φυσικά δικαιώματα τα οποία είναι απαράγραπτα και αδιέρετα. Και η χρήση των PNR θα μπορούσε να θίξει τα θεμελιώδη δικαιώματα, επομένως θα πρέπει να δράσουμε με την ίδια προσοχή και επιφυλακτικότητα, όπως αναφέραμε και για την περίπτωση του SWIFT. Τρίτη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω, ως γενική σκέψη, εγώ πιστεύω ότι η ασφάλεια και η ελευθερία δεν είναι δύο αρχές που αλληλοποκλείονται. Δεν είναι ένα παίγνιο μηδενικού αθρίσματος. Και όταν έχουμε περισσότερη ασφάλεια αυτό διαβρώνει αντίστοιχα την ελευθερία. Ή αν προστατεύουμε περισσότερα τις θεμελιώδεις ελευθερίες αυτό μειώνει την ασφάλεια αντιστοίχως. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα ψευδές δίλημα. Αντίθετα, νομίζω ότι η ασφάλεια και η ελευθερία είναι δύο αρχές οι οποίες ενισχύουν η μία την άλλη και οι δύο αυτές αρχές μπορούν να αναγνωριστούν και να ενισχύσουν η μία την άλλη ως αρχές που αποτελούν τμήμα των ε, συνταγμάτων, των βασικών νόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά έχουν ενσωματωθεί και οι δύο αυτές βασικές αρχές στην συνθήκη της Λισαβόνας. Από τη στιγμή που υπάρχει η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που εξασφαλίζει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτή η Χάρτα έχει ιερό χαρακτήρα και δεν μπορούμε να την παραβιάσουμε. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να σκεφτούμε και περισσότερο, πιο μακριά από το βραχυπρόθεσμο χρονικό πλαίσιο. Πρέπει να δούμε πιο μακροπρόθεσμα ποια θα ήταν τα μέτρα τα οποία θα εξασφαλίσουν την ασφάλειά μας, αλλά με το να εξασφαλίσουμε καταρχήν ότι τα μέτρα αυτά θα έχουν αποτελεσματικό χαρακτήρα και παράλληλα δεν θα θίγουν τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών γιατί αυτό είναι ένα στοιχείο και της ευμάρειας αλλά και της ίδιας ασφάλειας των πολιτών μας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η κυρία Μάλστρομ, για να κλείσει αυτή η συζήτηση ε, εξ ονόματος της Κομισιόν. Ε, φαντάζομαι θα έχετε δει περισσότερο από εσά το Minority Report, έκθεση της μειοψηφία. Ε, είναι ένα φοβιστερό φιλμ. Αυτή η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και επικοδομητική και γνωρίζω τις ομοιότητες με τη συζήτηση για το SWIFT, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και το θέμα της προστασίας ιδιωτικής σφαίρας των πολιτών. Ε, επικρίσεις για την προστασία των δεδομένων, διευκρινής των ε, στόχων, αβεβαιότητες κτλ. Οι διαπραγματεύσεις ε, επίσης μας, ε, που έχουν γίνει για το SWIFT μπορούν να μας εμπνεύσουν ε, για τα θέματα του PNR και νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει και τις ιδέες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τρία θεσμικά όργανα έχουν δουλέψει για αυτά τα θέματα, το Κοινοβούλιο, η Κομισιόν και το Συμβούλιο, μπορούν να συνεργαστούν για, για αυτά τα πολύ ευαίσθητα και λεπτά θέματα. Ελπίζω να υπάρξουν καλά αποτελέσματα. Άκουσα με προσοχή τη συζήτηση, διάβασα το ψηφισμά σας, είναι ισορροπημένο, συνετό και θα αρχίσουμε τη δουλειά πολύ γρήγορα με βάση αυτό το ψήφισμα. Ε, όπως ξέρετε, έχω υποσχεθεί στο Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της ακρόασής μου ότι θα κοιτάξω όλα τα μέτρα καταπολέμησης της τρομοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έχω μια συνολική γνώση και θα τα συζητήσω με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα συζητήσω τη συνολική στρατηγική μας για τον επιμερισμό των δεδομένων κτλ. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό και θα αυξηθεί η διαφάνεια. Σας ευχαριστώ λοιπόν ε, κυρία Πρόεδρε ε, σας ευχαριστώ και σας κυρίες και κύριοι βουλευτές. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την συνεργασία σας. Κλείνουμε λοιπόν τη συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει ε, στην πρώτη Ολομέλεια του Μαΐου.